<laughs> Γεια. Λοιπόν, καλώ ήρθατε στην Επιτροπή ε, Συνταγματικών Υποθέσεων. In den letzten sieben Jahren. μας τα τελευταία 7 χρόνια ουσιαστικά συνίστατο στο να καταλήξουμε σε μια νέα ε, μεταρρυθμιστική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως ξέρετε την ιστορία της συνθήκης αυτής και εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να ακούσουμε πως η τσεχική προεδρία βλέπει τα πράγματα τι εξελίξεις πρέπει να περιμένουμε του επόμενους μήνες το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο το Δεκέμβρη πήρε κάποιες αποφάσεις και ε, αναμένεται μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 να έχει περατωθεί η, συνθήκη, διαδικασία κύρωσης της συνθήκης. Υπάρχουν ε, επίσης αποφάσεις για τη μεταβατική περίοδο, για την ε, σύσταση κάποιων θεσμικών οργάνων ο αριθμός των ευρωβουλευτών είπε το Συμβούλιο κάτι για τον αριθμό των ευρωβουλευτών για τον διορισμό του Προέδρου της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όρισε και ορισμένα πράγματα για την Προεδρία του Συμβουλίου, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για το Συμβούλιο Υπουργών κτλ. Υπάρχει μια σειρά νομικών θεμάτων και πολιτικών θεμάτων προφανώς που μας ανησυχούν και γι' αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Εγώ έχω μια θητεία 10 ετών ουσιαστικά εδώ σε τούτο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε ε, και έχω περα, περάσει διάφορες προεδρίες ε, η Τσεχική Προεδρία είναι κάπως ιδιαίτερη βεβαίως είναι το πρώτο, η πρώτη χώρα του Συμφώνου της Βαρσοβίας που αναλαμβάνει την Προεδρία ε, και ε, γι' αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό η Προεδρία σας να στεφθεί από επιτυχία. Επίσης όμως θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν και κάποιοι δισταγμοί, κάποιοι σκεπτικισμοί οι οποίοι μας έρχονται από την τεχική δημοκρατία εκπλήσωμε από κάποια πράγματα που φαίνεται ότι λέγονται στη Γερουσία ξέρω ότι δεν είστε υπεύθυνους εσείς βεβαίως θα θέλαμε βεβαίως η κύρωση και η επικύρωση στη χώρα σας να είχε γίνει πριν από την ανάληψη της Προεδρίας για να ε, είστε ελεύθεροι να αγωνιστείτε για άλλα θέματα τώρα βέβαια τα πράγματα δεν έγιναν έτσι πρέπει πρώτα να τελειώσει η διαδικασία κύρωση στη χώρα σας πρέπει ακόμη μάλλον να τελειώσει διάβασα τι λέγεται στα ΜΜΕ με ξέπληξε κάποια πράγματα γιατί ε, ουσιαστικά τίθενται όροι και προϋποθέσεις για την ε, κύρωση μα όταν υπογράφεται μια συνθήκη από ένα κράτος μέλος ε, υπο, θέτω ότι είναι υποχρέωση του κράτους μέλους αυτού να ε, κυρώσει και όλα τελικά ε, την συνθήκη αυτή. Επίσης ε, Ακούσαμε ε, για τη Βαρσοβία ότι ε, πρέπει να περιμένουν μέχρι ότου να γίνει η κύρωση κάποια άλλη χώρα κτλ. Μα αν αρχίσουμε αυτό το παιχνίδι, το ότι περιμένω μέχρι ότου υπογράψει ή κυρώσει ο διπλανός μου, ο τον μου, φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Είναι λίγο ανοησία, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να ξεκινήσει ένα τέτοιο παιχνίδι, λέω εγώ. Εν πάση περιπτώσει στην Επιτροπή μας εκτός από αυτά τα σημαντικά θέματα έχουμε και άλλα θέματα ίσως λιγότερο σημαντικά αλλά ίσον σημασία ε, για την γενική πολιτική σκηνή αλλά αρκετά σημαντικά για μας έχουμε τις ομάδες πίεσης, ε, λόμπι που πιέζουν για ορισμένα πράγματα. Έχουμε το θέμα των agencies ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα ε, δημιουργηθούν, πώς θα ελεγχθούν. Το Κοινοβουλίο ανέκαθεν υποστήριζε ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη τάξη και αυστηρότερη όρη για τις υπηρεσίες αυτές. Ε, έχουμε επίκυνται οι, οι εκλογές και καλό θα ήταν να ξέρουμε τι θέλει και η Προεδρία και τι γίνεται και πώς ενημερώνονται οι πολίτες, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι κάνει το Συμβούλιο. Αλλά αρκετά μίλησα. Έχετε κυρία Αντιπρόεδρε το λόγο. Yeah, thank you, thank you very much, uh, Joe. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω καλημέρα σε όλους. Κάποιους ε, σας ξέρω από τις επαφές που είχαμε τις τελευταίους μήνες όταν ε, προετοιμάζαμε την Προεδρία μας αρκετά μεγάλη ευθύνη γιατί για μας είναι Μεγάλη υπόθεση, πρώτη φορά αναλαμβάνουμε. Προεδρία είναι το βάπτισμα του πυρός. Σε μια δύσκολη μάλιστα εποχή και διεθνές περιβάλλον. Οπότε ο στόχος μας, ο στόχος σημερινής μας ε, συνάντησης είναι να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της ε, Τσεχικής Προεδρίας για τους ε, επόμενους μήνες όπως είναι η παράδοση ξέρετε παρελάβουν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου όλοι σχεδόν η κυβέρνηση της Τσεχίας ε, ήρθε στις Βρυξέλλες για να παρα... να παραστείς διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οπότε συχνά η δεύτερη τρίτη εβδομάδα της Προεδρίας ήταν απλά η αρχή. Αλλά εμείς ξεκινήσαμε ήδη νωρίς νωρίς ε, την πρωτοχρονιά. Δεν προλάβα καλά καλά να γιορτάσω γιατί περιμέναμε τις δύο κρίσεις. Μία η Γάζα γιατί ήταν σε δύο φάσεις. Μία ήταν ε, οι βομβαρδισμοί τέλος Δεκεμβρίου και μετά είχαμε τη χερσαία εισβολή 3 Ιανουαρίου νομίζω Σάββατο βράδυ και μετά υπήρχε το φυσικό αέριο όπου είχαμε τις δατικές ε, επαφές και με τις δύο πλευρές οφείλω να πω πως ε, τουλάχιστον κάποιος μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης ε, που είχαμε συμφωνήσει πριν από τρία χρόνια με την ίδια πάλι κρίση λειτουργήσε Λάβαμε μια επιστολή από τον πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Γκασπρομ ε, και από τον αντιπρόεδρο της ε, ρωσικής κυβέρνησης λίγες μέρες πριν ότι θα έχουμε κάποια προβλήματα. Αλλά δεν περιμέναμε τόσα προβλήματα. Ίσως μία μείωση 40% ε, για δύο μέρες που είχαμε δει στο παρελθόν, αλλά κανείς δεν περίμενε τόσο ριζοσπαστικές κινήσεις να κόψουν τελείως το φυσικό αέριο στην Ευρώπη και να μείνει μισή Ευρώπη ε, να μπλεχτεί στο πρόβλημα. Κοιτάξτε, εμεί ε, προετοιμάζαμε το πρόγραμμά μας, μιλούσαμε για τα τρία ή που λέμε στα αγγλικά οικονομία, ενέργεια και νομίζω πως ήταν ένα από τα σημαντικότερα θέματα και όλες η ενέργεια για το Συμβουλίο του Μαρτίου και το τρέτο βεβαίως είναι είναι η Ευρώπη στον κόσμο και υπήρχε βεβαίως και η ανάγκη αλληλεγγύης εντός της Ευρώπης. Ωραία λόγια αυτά, αλλά όταν αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα και την ε, κατάσταση που έχουμε ότι δηλαδή έχουμε χώρες όπως Σλοβακία, Βουλγαρία και η Ουγγαρία ως ένα βαθμό τότε το ζήτημα εκεί το ζήτημα του φυσικού αερίου ήταν το πρώτο πολιτικό πρόβλημα, ήταν και το πρωτοσέλιδο. Ενώ βεβαίω αλλού στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο ήταν στις μέσα σελίδες των εφημερίδων. Οπότε για να διατηρηθεί η ενότητα της Ένωσης ε, και να μπορεί να δρά αποτελεσματικά αλλά και για να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε την Ένωση κατά τρόπον ώστε να μην ε, δημιουργήσουμε άλλο πρόβλημα γιατί το θέμα ήταν ποιος ε, ποιος έφταιγε σε ποιον θα θα έπεφτε το, το φταίξιμο για να μην καταλήξουμε εμείς να πληρώσουμε τα σφάλματα των άλλων. Ε, η αρχή λοιπόν ήταν δύσκολη, αλλά τα καταφέραμε. Πρώτα απ' όλα πιέσαμε και τους Ουκρανούς και τους Ρώσους να κάτσουν σε ένα τραπέζι, γιατί ε, ούτε να διαπραγματευτούν δεν ήθελαν και καταφέραμε χάρη στην συμφωνία παρατηρητών, να στείλουμε παρατηρητές δηλαδή στις, ε, στους αγωγούς και να κάτσουν να συζητήσουν και μετά καταφέραμε να αποφύγουμε το διχασμό της ε, Ευρώπης γιατί οι Ρώσοι προσκαλούσαν ε, τους καταναλωτές του αερίου τους σε μια προσπάθεια να μας διχάσουν και δεν ήταν εύκολο να πείσουμε κυρίως τους κορυφαίους πολιτικούς στην Πρατσλάβα, Σόφια και αλλού να βασιστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εδώ για να βοηθήσει. Οφείλουμε λοιπόν να αντλήσουμε το δίδαγμα ότι η αλληλεγγύη την οποία συχνά επικαλούμαστε μέσω πρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα έπρεπε να μετατραπεί σε πραγματικά, σε ουσιαστικά μέτρα. Στην περίπτωση στην οποία κινδυνεύουν τα ζωτικά συμφέροντα κάποιων κρατών μελών. Με συγχωρείτε για αυτή την εισαγωγή. Αρχικά μου είπαν να κάνω μια γενική εισαγωγή 5 λεπτών για το πρόγραμμα. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ ενδιαφέρει να πω λίγα λόγια για το τι ε, έχουμε ήδη κάνει στις ε, τρεις πρώτες ε, εβδομάδες της Προεδρίας μας, αν και δεν αφορά άμεσα την Επιτροπή τη δική σας των συνταγματικών υποθέσεων. Ποιο είναι τώρα το θέμα της συζήτησής μας. Λοιπόν, εάν δούμε την Προεδρία που έρχεται εγώ θα την χώριζα σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά ζητήματα οικονομίας ενέργειας και κάποια εξωτερικών υποθέσεων. και θα έχουμε και το αποτέλεσμα του Συμβουλίου του Μαρτίου και μετά έχουμε το δεύτερο μισό, αν θέλετε, το δεύτερο τρίμηνο που θα είναι εξίσου σημαντικό από πλευράς θεσμικής γιατί θα προετοιμάζεται το Ευρωκοινοβούλιο για ευρωεκλογέ και θα προετοιμάζουμε και το Συμβούλιο του Ιωνίου που θα λάβει κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Θα έχουμε πρώτα απ' όλα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Έχουμε νομίζω παραδείγματο χάρη την υποχρέωση που αναφέρεται σαφώς στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου και αφορά τον ε, ορισμό του μελλοντικού πρόεδρου της Κομισιόν, μελλοντός πρόεδρου της και μετά έχουμε και τη συνθήκη της Λισαβόνας που επίσης αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Εδώ πέρα οπωσδήποτε καλωσορίζουμε τη συμφωνία που επιτευχθεί στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου για το τι πρέπει να γίνει από εδώ με την συνθήκη της Λισαβόνας και ευχαριστούμε και την Γαλλική Προεδρία για το ότι πέτυχε αυτή τη συμφωνία αλλά και την Ιρλανδική κυβέρνηση Θεωρούμε πως ε, το αποτέλεσμα αυτό είναι ισορροπημένο. Μετά από έτοιμα της Ιρλανδίας ε, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν πως θα δώσουν κάποιες νομικές εγγυήσεις για ζητήματα τα οποία αποτελούσαν πηγή ανησυχίας ε, στο δημοψήφισμα το περσινό στην Ιρλανδία. Και μετά ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για αυτά τα ζητήματα για να υπάρξει κάποια επιτυχής κατάληξη και δεσμεύτηκε άρα και η Ιρλανδική κυβέρνηση πως θα προσπαθήσει να ακυρώσει την συνθήκη μέχρι το τέλος της θητείας αυτής της Κομισιόν. Οι διάλλες κυβερνήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν ανάλογες προσπάθειες. Το ΔΕ Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είπε πως θα ληφθεί υπόψη η καθυστέρηση διαδικασία αυτή της επικύρωσης. Άρα συγκεκριμένα προβλέπονται μεταβατικές ε, διατάξεις ε, για την οργάνωση της ε, Προεδρίας που θα ακολουθήσουν τη θέση σε ισχύ της συνθήκης και κάποιες άλλες ρυθμίσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη 2009-2013. Το αποτέλεσμα βεβαίως αυτό είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας και οπωσδήποτε χρειάζεται να κάνουμε και άλλα πράγματα για τι μελλοντικέ ε, νομικέ εγγυήσεις και συμφωνήσαμε τον Δεκέμβριο πω αυτό θα γίνει μέχρι τα μέσα του 2009, δηλαδή μέχρι το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό του Ιουνίου. Γι' αυτό εμεί θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να γίνει σεβαστή αυτή η ημερομηνία. Για να τελειώσουμε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω δύο τομείς που αφορούν ιδιαίτερα την Προεδρία μας ε, σε σχέση με τις συνθήκες Λισαβόνας. Πρώτον, ο ενισχυμένος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο βεβαίω σημαίνει μεγαλύτερη δημοκρατία και λογοδοσία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και οπωσδήποτε η έμφαση στην περισσότερη επικουρικότητα και τον δημοκρατικό έλεγχο θα φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς πλησιάζει και η προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογέ. Οπότε οπωσδήποτε παρακολουθούμε από κοντά τις απόψεις της Επιτροπής σας που τους ανέφεραν ο Τζο Λάινεν, ο Έλμαρ Μπρόκ και την έκθεση Δεάν και λοιπόν ρωτήσατε για τη χώρα μου, Είδε δε στο κοινοβούλιο μας συνεχίζεται. Είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση χθε στην Επιτροπή Εξωτερικών. Νομίζω πως θα γίνει άλλη μια συνεδρίαση κάποιων σημαντικών επιτροπών ε, αρχές Φεβρουαρίου γιατί υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και μετά θα έχουμε την ψηφοφορία στην Ολομέλεια για δύο ζητήματα. Πρώτον, την ίδια τη συνθήκη της Λισαβόνας και δεύτερον, η δεσμευτική εντολή για, την απλο... για τις απλοποιημένες διατάξεις τροποποίησης της ε, συνθήκης κατά το οποίο θέτησαν ορισμένα κράτη-μέλη όπως ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία, Φιλανδία, τουλάχιστον αυτό ε, ξέρω εγώ. Και μετά οπωσδήποτε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οπότε η κυβέρνηση σκοπεύει να μας οδηγήσει αυτό το επιτυχές αποτέλεσμα. Και επιτυχία βεβαίως σημαίνει πως η ποιότητα εδώ προέχει της ε, ταχύτητας γιατί η ταχύτητα ορισμένες φορές μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Και βεβαίως δεν το θέμα αυτό. Να πω τώρα λίγα λόγια για κάποιο ένα ζήτημα, για κάποιο άλλο ζήτημα το οποίο απασχόλησε και την Επιτροπή Ελευθεριών πριν από λίγες ημέρες και αφορά την διαφάνεια θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια συμπεράσματα που έβγαλε το Συμβούλιο από την πρακτική του εμπειρία με την εφαρμογή του κανονισμού 1049 και να σχολιάσω και λίγο κάποιες από τις αναγκές αναθεώρησης του σημαντικού αυτού νομοθετικού μέσου. Οπωσδήποτε γνωρίζει το Συμβούλιο πως χρειάζεται κάποια επικαιροποίησει αυτός ο κανονισμός, αλλά παραμένει πεπισμένο το Συμβούλιο πως συνολικά λειτουργεί πολύ καλά αυτός ο κανονισμός και η εφαρμογή του δεν έχει δημιουργήσει μεγάλες δυσκολίες από όταν τέθη ενισχύ το Δεκέμβριο του 2001. Η ύπαρξη ενός κεντρικού αρχείου εγγράφων που είχε ήδη γίνει πριν τεθεί ενισχύ ο κανονισμός προφανώς έπαιξε ένα ρόλο. Τα δημόσια αρχεία των ε, εγγράφων του Συμβουλίου που περιέχουν πάνω από ένα εκατομμύρια έγγραφα από το 1999 και μετά τροφοδοτείται από ένα ηλεκτρονικό σύστημα το λεγόμενο workflow. Δεν θέλω τώρα να πω λεπτομέρειες γιατί οπωσδήποτε εσείς ε, θέλετε να συζητήσουμε και αν ε, σας ενδιαφέρει μπορούμε να επανέλθουμε. Σε γενικές γραμμές νομίζω πως ε, θα συνεργαστούμε μαζί σας και είναι λίγο νωρίς αυτή τη στιγμή να σχολιάσουμε λεπτομερώς ε, κάποιες προτάσεις που έγιναν από τις επιτροπές του Κοινοβουλίου και πρέπει τώρα να ενσωματωθούν στην τελική έκθεση για την οποία είναι αρμόδια η Επιτροπή Ελευθεριών. Καλό θα ήταν λοιπόν να γνωρίζουμε πως το υπάρχον καθεστώς πρόσβαση για Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν χαρακτηρίζεται από κάποια άλλα πράγματα. Ε, π.χ. στο μέλλον θα διευρυνθεί το δικαίωμα πρόσβασης και ο ορισμός του εγγράφου και η, δυνατότητα των και η υποχρέωση των θεσμικών οργάνων να εξτάζουν κατά περίπτωση τα έγγραφα που ζητάει το κοινό με βάση το λεγόμενο, το λεγόμενο τεστ βλάβης. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποια είναι η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην προστασία κάποιων προσωπικών και ιδιωτικών σφαιρόντων και την πρόσβαση του κοινού τρίτο θέμα που μπορεί να, να σας ενδιαφέρει είναι αυτό που λέμε Europe in Partnership πολύ ενδιαφέρον θέμα ιδιαίτερα εν ώψη των ευρωεκλογών ε, και μεγάλη πρόκληση βέβαια και για το Συμβουλίο και για τα κράτη-μέλη. Όπως θα θυμάστε τέλη Οκτωβρίου πέρσι το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβουλίο έκαναν ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά και ε, ε, γιατί ε, ξέδωσαν ουσιαστικά την ανακοίνωση αυτή, μάλλον την πολιτική δήλωση με τίτλο European Partnership, όπου λένε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η, το θέμα σε όλα τα κράτη-μέλη των σχέσεων με το, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και με τους ε, άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Όπως ξέρετε έχουμε πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε τις ευρωεκλογέ από τη μια, τις κλιματικές αλλαγές από την άλλη και το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ παίζουν και Αμερικανοί και άλλοι σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι βεβαίως και η επέτειος της κατάρρευσης του σιδηρού παραπετάσματος λέει ο, μιλητή, στην Ευρώπη και την επέτειο αυτή θα την ε, γιορτάσουμε φέτος. Επίσης είναι η απάντηση της ε, Ευρώπης στην χρηματοπιστωτική κρίση στην, και στην οικονομική ύφαση. Ε, ειδικά σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Σε ό,τι αφορά τη, τις εκλογές του 2009, οι ευρωεκλογέ μας δίνουν μια καλή ευκαιρία για να ενδυναμώσουμε την επικοινωνία με τους πολίτες για κάποια θέματα και για να υπάρξει μια εταιρική σχέση ε, με τους πολίτες για τα πολιτικά θέματα. Θέλουμε λοιπόν να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο και το Κομισιόν για αυτόν τον λόγο για να εφαρμόσουμε επιτυχώς την ε, στρατηγική που αναφέρει η ε, ανακοίνωση. Θα ήθελα εν παρόδο να υπενθυμίσω ότι η τσεχική κυβέρνηση ε, προωθεί τα θέματα τα, της δημοκρατικής αλλαγής επ' ευκαιρία της 20ης επαιτίου της έλευσης της δημοκρατίας. Θέλουμε να γιορτάσουμε ε, μια πολύ σημαντική αλλαγή στην ευρωπαϊκή ιστορία, να προωθήσουμε τις ουσιαστικές ελευθερίες, το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και όλες τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ευρώπη. Θα ήταν χρήσιμο, ειδικά για εκείνους που δεν ε, είχαν την εμπειρία από πρώτο χέρι να ζήσουν αυτά γεγονότα και δεν έζησαν αυτά γεγονότα, ε, να καταλάβουν ότι οι αξίες τις οποίες απολαμβάνουμε τώρα δεν είναι αυτονόητες και δεν υπήρχαν πάντα. Προφανώς η Προεδρία θα ήθελε να συνεργαστεί και με άλλα θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά τις ενημερωτικές εκστρατείες για άλλα σημαντικά θέματα, ενέργεια, κλιματικές αλλαγές ε, και χρηματοπιστωτική κρίση φυσικά. Τελευταίο σημείο για τις ρυθμιστικές υπηρεσίες η ομάδα εργασίας εξέτασε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους ευρωπαϊκούς αυτούς οργανισμούς, όπου προτείνεται η έναρξη ενός διαθεσμικού διαλόγου για να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση για αυτές τις υπηρεσίες. Στις 30 Νοεμβρίου το Συμβούλιο απάντησε θετικά στην πρόσκληση που έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής στις 7 Μαΐου του 2008 για να συμμετάσχει στην διαθεσμική ομάδα εργασίας με σκοπό να συζητηθεί η κοινή προσέγγιση για αυτές τις ρυθμιστικές, ε, τους ρυθμιστικούς οργανισμούς. Ε, ένα αντίγραφο της επιστολής στάληκε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του κύριου, τον κύριο Πέτερη. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο των υπηρεσιών αυτών για την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών και συμμερίζεται το μέλημα ότι πρέπει να γίνουν πολύ πιο αποτελεσματικό εργαλείο. Επομένως, είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε μαζί με την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία και τη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών, αυτών των οργανισμών. Θέλουμε λοιπόν να γίνει η πρώτη συνεδρίαση, περιμένουμε με υπομονησία την πρώτη συνεδρίαση του διαθεσμικού αυτού, α, της διαθεσμικής ομάδας εργασίας που θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στο Φεβρουάριο. Εν κατακλείδη, κύριοι βουλευτές, σας ανέφερα κάποια θέματα, δεν τα εξάντλησα όμως, ε, ούτε μίλησα πολύ για την επιτροπολογία, ούτε για τις ευθύνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, ούτε για τα εθνικά κοινοβούλια υπό τη νέα συνθήκη. Φυσικά έχουμε χρόνο, τα συζητήσουμε όλα αυτά με περισσότερες ε, λεπτομέρειες είχε προβλεφθεί ούτω ή ένα χρονικό διάστημα 45 λεπτών για κάτι τέτοιο. Σα ευχαριστώ. So, Alexander thank you very much for... Ευχαριστώ, κύριε Βόντρα, που μας παρουσιάσατε κάποια σημαντικά θέματα που θα απασχολήσουν την Τσεχική Προεδρία. Την πρωτοχρονιά εξάλλου, από την πρωτοχρονιά άρχισε να φαίνεται το νέο κλίμα. Ε, η πρώτη και η δεύτερη κρίση ε, με τη Γάζα καταρχήν, που σας επηρέασαν. Και μετά το φυσικό αέριο. Και τα δύο αυτά θέματα συνδέονται με την μεταρρυθμιστική συνθήκη. Ξέρετε ότι η αλληλεγγύη είναι μία από τις αρχές που είναι εγγεγραμμένη στη νέα συνθήκη. Και η ενεργειακή πολιτική για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια θα είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, Διάφοροι πολιτικοί από την Ευρώπη συνέρευσαν εκεί. Ο Κουσνέρ, Σολάνα, ο Σαρκοζή, ο Στάινμάγερ. Κανένας όμως ε, δεν παίρνει την Ευρώπη στα σοβαρά. Ο καθένας λέει τα δικά του. Ένας εκπρόσωπος με μεγαλύτερο ρόλο με βάση τη νέα συνθήκη θα μπορούσε να είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου που θα μιλήσω με, μία φωνή, με, μία συγκεκριμένη φωνή και θα εκφράζει όλη την Ευρώπη. Το να μιλάμε με μία φωνή λοιπόν είναι κάτι που θα μας το εξασφαλίσει η νέα συνθήκη και το χρειαζόμαστε αυτό. Μιλήσατε επίσης κύριε Βόντρα για τις εγγύησει που οι εταίροι πρέπει να δώσουν στην Ιρλανδία Βέβαια πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτός ο όρος εγγύηση, εγγύησης. Θεωρώ ότι κάποια από τα σημεία είναι προφανή. Η φορολογική πολιτική αποφασίζεται ομόφωνα. Τι περισσότερες εγγυήσεις χρειάζεται κάποιος. Δεν νομίζω ότι στην πολιτική μπορεί κανείς να δίνει αιώνιες εγγύησεις. Ότι ποτέ στο μέλλον τίποτα δεν θα αλλάξει μια τέτοια εγγύηση δεν μπορεί να τη δώσει κανένας. Χθε, διάβασα στο New Observer ένα άρθρο από ένα μέλος ε, της ε, Γερουσίας που μιλούσε για αυτές τις ε, εγγυήσεις προς την Ιρλανδία που θα έπρεπε να είναι εγγύησεις και προς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και κυρίως βεβαίως και προς την Τσεχία. Μιλάμε για ένα Τσέχο γερουσιαστή. Δεν ξέρω αν εκφράζει όλους, τι ακριβώς σημαίνουν αυτά τα λόγια. Σας περιμένουν πολλοί ομιλητές που θα σας υποβάλουν ερωτήσεις. Ο κύριος Ντεχάν είναι ο πρώτος, που είναι και εισηγητής για την διαθεσμική ισορροπία για αυτή την έκθεση συγκεκριμένα. Ο κύριος Ντεχάν. Ε, eh, Ευχαριστώ την Τσεχική Προεδρία που μας δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε διάφορα πράγματα. Θα επικεντρωθώ στη μεταβατική περίοδο όπως ε, διαγράφηκε από τα, συμβούλια, από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Και κυρίως θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο σημεία. Καταρχάς, σε ένα σημείο που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς είπαμε ότι αυτή τη στιγμή στη συνθήκη της Λισαβόνας τεθεί σε ισχύ, διάφοροι βουλευτές σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στη συνθήκη της Λισαβόνας, ο αριθμός των βουλευτών θα αυξηθεί. Το θέμα είναι πώς θα εκλεγούν αυτοί οι βουλευτές. Είναι θέμα των κρατών μελών, των ενδιαφερομένων κρατών μελών να μεριμνήσουν για αυτό το θέμα. Και στην ενδιάμεση περίοδο τι θα γίνει με αυτά τα μέλη, τα νέα μέλη του Κοινοβουλίου όσο δεν υπάρχει δηλαδή πρωτόκολλο για να εγγυάται τις έδρες των βουλευτών. Νομίζω λοιπόν ότι τα κράτη θα έχουν κάποιες ιδέες για το πώς θα τους εκλέξουν, αλλά θα υπάρξει μια περίοδος αβεβαιότητας. Όσο η συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχει εγκριθεί, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι τίποτα γιατί η νομιμότητά τους προκύπτει από αυτή τη συνθήκη. Αλλά και αφού εγκριθεί η συνθήκη και όσο δεν υπάρχει το πρωτόκολλο θα έχουν εκλεγεί ιονοί ας πούμε. Και στην πραγματικότητα γίνονται ε, ευρωβουλευτές με όλα τα δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή στο συμπληρωματικό πρωτόκολλο ε, έχει συμπεριληφθεί στην ε, συνθήκη προσχώρησης των κρατών μελών. Αυτή είναι η ερμηνεία μου. Είναι σωστή αυτή η ερμηνεία. Δηλαδή, τα εθνικά κράτη θα αποφασίσουν πώς αυτά τα επιπλέον μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εκλεγούν και εν συνεχεία θα υπάρξει μία περίοδος αβεβαιότητας όσο δεν έχει εγκριθεί η συνθήκη της Λισαβόνας και αυτή τη στιγμή εγκριθεί η συνθήκη της Λισαβόνας θα είναι βουλευτές μεν αλλά ιονοί και θα γίνουν πραγματικά μέλη του Κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή υπάρχει το πρωτόκολλο. Εγώ τουλάχιστον έτσι ερμηνεύω τα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου. Ε, θα ήθελα να μου πείτε αν η ερμηνεία μου είναι σωστή. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερον, δεύτερο συμπέρασμα, πολύ σημαντικό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Λέμε, αμέσως μετά τις ε, ευρωπαϊκές εκλογές θα ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα προβεί στο διορισμό του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εδώ έχω κάποιες ερωτήσεις να σας θέσω. Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αμέσως μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές θα διέπεται από τη συνθήκη της Νίκαιας, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν διαφορέ ανάμεσα στη Νίκαια και στη Λισαβόνα σε ό,τι αφορά το διορισμό του Προέδρου τη ε, Κομισιόν. Στα πλαίσια τη Νίκαια, ο Πρόεδρο διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και επικυρώνεται αυτή η απόφαση από το Κοινοβούλιο, ενώ με βάση τη Λισαβόνα ε, αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει λοιπόν μια πρώτερη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν κάνει μια πρόταση το Συμβούλιο. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Η Τσεχική Προεδρία πώς θα προσεγγίσει αυτό το θέμα. Νομίζω ότι τουλάχιστον για το Κοινοβούλιο, αυτή είναι η πρότασή μου, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να πει ότι ακόμη και αν δεν εφαρμόζεται ακόμα η Λισαβόνα, η διαδικασία της διαβούλευσης θα πρέπει να ισχύσει και θα πρέπει να υπάρχει στη διάθεσή μας και ο κατάλληλος χρόνος. Νομίζω ότι στις 16 Ιουνίου θα γίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μου φαίνεται αδύνατο ανάμεσα στις εκλογές ε, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να γίνει μία διαβούλευση με τις πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Ε, δηλαδή η προθεσμία ανάμεσα στα δύο γεγονότα είναι πάρα πολύ βραχία. Η Προεδρία έχει την ε, πρόθεση να ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα. Και, και μια συμπληρωματική ερώτηση. Περιμένετε από το Κοινοβούλιο να επιλέξει τον πρόεδρο πριν να έχουμε την βεβαιότητα για τη Λισαβόνα ή ούτως ή άλλως. Και νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Αν προβλέψουμε ότι η Λισαβόνα θα επικυρωθεί, δεν έχει κανένα νόημα να αρχίσουμε την, να συνθέτουμε την Κομισιόν όσο παραμένει μια βεβαιότητα. Γιατί η σύνθεση της Κομισιόν και η παρουσία του εκπροσώπου της εξωτερικής πολιτικής του αντιπροέδρου γίνεται στα πλαίσια της Λισαβόνας. Αν εγκριθεί η Λισαβόνα, το Κοινοβούλιο θα πρέπει Θα πρέπει μάλλον να περιμένουμε να ε, επικυρωθεί η Λισαβόνα πριν περάσουμε στο διορισμό των μελών της Επιτροπής, για να το πω έτσι. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία. Συμφωνεί η Τσεχική Προεδρία με την ανάλυση μου. Τελευταία παρατήρηση, Πρόεδρε. Ερώτηση και πρόταση προς την Τσεχική Προεδρία. Θα έπρεπε η Προεδρία να έρθει σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε διαβούλευση αν θέλετε, πριν διαλυθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να δούμε πώς θα κινηθούμε μετά τις εκλογές. Γιατί αν δεν το κάνουμε και αν το νέο κοινοβούλιο αρχίσει να παίζει και να συνθέτει έτσι αυθαίρετα, δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και πρέπει να το παίξει πολύ γρήγορα. Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες ανάμεσα στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο στο νέο Κοινοβούλιο να, να ξέρει τι μέλη γενέστε. Ευχαριστούμε, Ζαν Ντεάν. Σημαντικά τα ερωτήματα. Πρέπει να κλείσω όμως το κατάλογο των ομιλητών γιατί ο χρόνος πιέζει. Ρίτσαρτ Κόρμπετ, λίγο πιο σύντομα. Είπα χτε πω πρώην πρωθυπουργοί μπορούν να μιλήσουν λίγο παραπάνω και οι συγητές βεβαίω. Οπότε έχετε τον λόγο. Ναι, εγώ μια σύντομη και απλή ερώτηση έχω στην ε, χώρα μου υπάρχει δυνατότητα να στοιχηματίζει κανείς και για πολιτικά γεγονότα. Πότε π.χ. θα γίνουν οι επόμενες εκλογές, πώς ε, θα είναι η πλειοψηφία των εργατικών μετά τις εκλογές. Σε τέλος πάντων για ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς στοιχηματίζουμε. Το ερώτημά μου είναι Εάν είναι να στοιχηματίσω πότε θα ακυρώσει τελικά η τσεχική κυβέρνηση τη συνθήκη της Λισαβόνας, ποια ημερομηνία θα με συμβουλεύατε να παίξω. Simple and short question. Okay. Uh, Enrique... Και σύντομο το ερώτημα. Ε, ε, Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω και εγώ με τα ερωτήματα του κυρίου Ντεάν. όσον αφορά την ε, σύνθεση του Κοινοβουλίου αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο τόνισε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 18 ευρωβουλευτές από 12 κρατημέλη που αναμένουν να τεθεί ισχύ αυτή η συνθήκη. Μιλάμε εδώ πέρα βεβαίως για το για την σύνθεση όπως είπα του Κοινοβουλίου και μετά υπάρχουν και οι νομοθετικές ε, εξουσίες που θα ασκήσουμε στο μέλλον. Το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο τη μία ή την άλλη χώρα, μας επηρεάζει όλους τώρα. Υπάρχουν κάποιοι ευρωβουλευτές που κατέθεσαν ε, μία τροπολογία στην ε, γνωμοδότηση Κόρμπετ για τον νέο κανονισμό Οπότε τα κράτη-μέλη τα οποία είναι στον κατάλογο μπορούν να θεωρούνται παρατηρητές μέχρι να κυρωθεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση, αλλά τέλος πάντων είναι μια λύση λειτουργική εν αναμονή της απόφασης άλλων κρατών μελών μεταξύ των οποίων και η Τσεχία. Σύμφωνα δε με τις πληροφορίες που έχω λάβει νομίζω πως υπάρχει άλλη μια αναβολή της ε, κύριας συνθήκης Λισαβόνας από το τσεχικό κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση η κυβέρνησή σας θεωρεί πως η συνθήκη αυτή πρέπει να παραμένει όμοιρος των εξελίξεων με την αντιπυραυλική ασπίδα. Αυτό είναι κάτι που επηρεάζει όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρνητικό τρόπο, οπότε θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποια είναι η επίσημη θέση της Τσεχίας. Σας ευχαριστώ, Άντριου Νταφ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά βλέπω εκπρόσωπο της Τσεχής Προεδρίας εδώ. Και το λέω αυτό γιατί εδώ και κάμποσο καιρό η Επιτροπή μας παρακολουθεί το τι συμβαίνει στην Τσεχία στο συνταγματικό επίπεδο. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω σχετικά. Δυο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω πρώτον. Είναι πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε για πολιτικούς ηγέτες, βασιλιάδες και βασίλισσες που ε, δεν κατάφεραν ε, ή δεν, έκαν, δεν εξετέλεσαν όπως έπρεπε τις εντολές των κοινοβουλίων τους. Ε, ο κύριος το Πολάνεκ στο Στρασβούργο είπε ότι θεωρεί την συνθήκη της νίκης καλύτερη από την μεταρρυθμιστική συνθήκη. Δεν ξέρω αν αυτό φίλε το, αυτό που είπε οφείλεται σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους Ιρλανδούς να υπερψηφίζουν τη συνθήκη δεν νομίζω αλλά είναι λίγο παρακινδυνευμένο να προσπαθήσει προσπαθεί ε, κανείς να μετατρέψει κάποια από πολιτική άποψη απλά πράγματα σε νομικές εγγυήσει που υπόσχεται κανείς. Είναι και είναι και δύσκολο να το κάνει κανείς αυτό. Έχω ένα ερώτημα σχετικά με την υπόθεση του Προέδρου Σαρκοσί ότι το ότι η δέσμη μέτρων που έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει τους Ιρλανδούς μπορεί να συναρτηθεί με την να ή μάλλον να ε, να μαζί και να προσαρτηθεί στο, στην πράξη προσχώρησης της Κροατίας. Ή αυτό ε, φαντάζομαι ότι δεν Δεν θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Τσεχικής Προεδρίας και την γνώμη που έχετε για τη θέση του κυρίου Σαρκοζή. Και αν υποστηρίζετε τέλος πάντων αυτή την ιδιαίτερα ε, αυθάδη ε, δήλωση που έκανε ο πρόεδρος Σαρκοζή στο τέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Ναι, λέει ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ, καλά κάνετε και θέσατε το θέμα της δήλωση του Πρωθυπουργού το Πολάνεξ στο Στρασβούργο. Είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε κάποιες διευκρινήσεις σχετικά. Τώρα, ε, ε, είδα ε, κάτι στον τύπο που έλεγε ότι ε, πολλά μέλη του, της Γερουσίας ε, προτιμούν τη συνθήκη της νίκης γιατί θεωρούν πιο δημοκρατική από τη συνθήκη της Λισαβόνας εγώ θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο αλλά τέλος πάντων τι μου well, sadly, Πρόεδρε δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα Ξεκινώντας την παρέμβασή μου δηλώνω σαφώς ότι το θέμα της συνθήκης είναι σαφώς θέμα τσεχικό, θέμα της Τσεχίας, της Τσεχικής Βουλής και των πολιτικών ηγετών της χώρας. Από εκεί και πέρα η Τσεχία λοιπόν αποφασίζει τι θα κάνουμε τη συνθήκη και δεν μπορούμε να προσπαθούμε εμεί να επιβάλλουμε πράγματα στη χώρα αυτή. Πρόκειται για μια δημοκρατική χώρα με μακρά ιστορία και οι δημοκρατικοί θεσμοί της χώρας αυτής είμαι πεπισμένος ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση στο τέλος πάντως περιμένω με ενδιαφέρον να δω τα αποτελέσματα εγώ στην παρέμβασή μου θα ήθελα να πω πρώτον ότι με ενθαρρύνει ιδιαίτερα με ενθαρρύνει ιδιαίτερα αυτά που είπε ο κύριος Τοπολάνεξ στο Στρασβούργο ο οποίος πρότεινε και ένα πολύ καλό πρόγραμμα για την τσεχική προεδρία. Ε, ο κύριος Βόντρα επανέλαβε ορισμένα πράγματα σήμερα. Το θέμα της ασφα... ενεργειακής ασφάλειας είναι ζωτική σημασία κατά την άποψή μου και αν η τσεχική δημοκρατία καταφέρει να καθησυχάσει τους φόβους και τις ανησυχίες μας για το θέμα αυτό. Αυτό και μόνο θα ήταν πραγματικό κατόρθωμα. Θα ήθελα, μια και είναι ο κύριος Βόντρα εδώ, ε, θα ήθελα να μας πει ε, κάποιες παρατηρήσεις που έγιναν από τον τύπο, από τα μίντια για τε, κάποιες αμφιβολίες που ακούστηκαν για το κατά πόσο η Τσεκή Προεδρία θα επιτύχει βεβαίως. Η Γαλλική Προεδρία προηγήθηκε. Οι Σουηδοί ακολουθούν. Όντως η Τσέχικη Προεδρία είναι, βρίσκεται σε ένα λαβά, ε, ε ενία σε μια ε, παράξενη χρονική στιγμή αλλά έχει τους πόρους η Τσεχία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της Προεδρίας ε, και βεβαίως η Ευρώπη τελικά θα πάρει τις αποφάσεις αλλά ο κύριος Φόντρα θα ήθελα να ξέρω αν πιστεύει ότι μπορεί πράγματι μια μικρή χώρα να κάνει μια επιτυχή προεδρία βεβαίως συντονισμός, επικαλύψεις, βοήθεια ιδιαίτερα από τους, από τους Γάλλους υπήρξε και οι Σουηδοί το ίδιο προσπαθούν να βοηθήσουν για να προετοιμάσουν και τη δική τους προεδρία ε, αυτού του είδους η βοήθεια ή η στήριξη είναι καλή για την τσεχική προεδρία. Και κάτι τι άλλο για τη διαφάνεια. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ε, ζητούμε να είναι δημόσιες συνεδριάσεις του Συμβουλίου ούτως ώστε η γνώμη να ξέρει τι γίνεται στο Συμβουλίο εξ ονόματός της. Η Τσεχική Προεδρία τι πιστεύει η Βρετανική κυβέρνηση εντωμεταξύ λέει ότι ε, τελικά ε, κατάφερε να επιτύχει πλήρη διαφάνεια στο Συμβούλιο. Αυτό δεν το πιστεύω εγώ. Ο κ. Βόντρα τι πιστεύει. Από εκεί και πέρα βεβαίω εμεί θέλουμε οι πολίτες να ενδιαφέρονται για την Ευρώπη και να προσέλθουν μαζικά στις ευρωεκλογέ. Η Προεδρία έχει κάτι κατά νου που θα μπορούσε να κάνει. Ε, πρόκειται να αναλάβει καμιά πρωτοβουλία γιατί ακριβώς ε, έχει την Προεδρία σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή όταν επίκυνται τον Ιουνίου ευρωεκλογέ. Πρόεδρος, ευχαριστώ απλώς λέω ότι θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Έκλεισα μάλλον. Έχετε το λόγο. Κάρλος Κανέρο, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους. Είμαι σίγουρος πως η Τσεχική Προεδρία με τις ε, δραστηριότητες της ε, θα κάνει αυτά τα οποία ζήτησαν οι συνάδελφοι, δηλαδή θα δημιουργήσει μια πιο ισχυρή Ευρώπη και είναι σαφές πως ε, πρέπει να ενισχύσουμε τα θεσμικά όργανα της ε, κοινότητας ε, για να μην διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Τώρα ένα ερώτημα. Ο κύριος Τοπολάνεκ όταν ήρθε στο Στρασβούργο είπε κάτι το οποίο φάνηκε δυσάρεστο στον Άνδριο, δηλαδή ότι ε, δεν ε, συμφωνούσε απολύτως με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θεωρεί η τσεχική κυβέρνηση ότι η, κυβέρνηση, η συνθήκη με ήταν καλύτερη συνθήκη. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ανακούφιση να ακούμε μια φορά μια ρεαλιστική και προσγειωμένη ανάλυση των προβλημάτων που κληρονομήσαμε και έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα έτσι ενός ε, όψιμου Ναπολέοντα ο οποίος κυκλοφορεί στην Ευρώπη και κατεβάζει σημαίες και ανεμίζει μόνο την ευρωπαϊκή σημαία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την ε, προσέγγιση σας. Δεν θα σας διέφυγε ασφαλώς η ηρωνία το ότι ο πρόεδρος αυτής της Επιτροπής αλλά και του Κοινοβουλίου κάνουν μάθημα στην τσεχική δημοκρατία για το ότι η Λισαβόνα πρέπει να κυρωθεί όταν η ίδια τους η χώρα ακόμα δεν έχει επικυρώσει τη συνθήκη. Εγώ ήμουν στην Πράγα, θα θυμάστε με την Επιτροπή αυτή, όταν σας επισκεφτήκαμε. Και άκουσα μετά για την ε, επίθεση που δέχτηκε ο πρόεδρός σας στην ε, επίσκεψη, στην συνάντηση που είχα μαζί του και ελπίζω να γνωρίζετε τώρα πια πως έχετε αρκετούς υποστηρικτές σε αυτό το κοινοβούλιο που θεωρούν ότι πρέπει να επιμείνετε στις θέσεις σας, ε, αντισταθείτε και να κάνετε ό,τι θεωρείτε σωστό κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Mr. Κύριος Βιλαβιεύσκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης που μας τονίσατε την αυξανόμενη σημασία του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά πρέπει να σας πω ότι από τις εθνικές μου εμπειρίες είμαι αρκετά απεσιόδοξος. Μετά το 2004, μετά την ένταξή μας, ε, επί δύο-τρία χρόνια ε, φτάναν σε εμά διάφορα σχέδια στην Επιτροπή μας, τα οποία πρέπει να εξετάσουμε. Το θέμα είναι από συνταγματικής απόψης, να δούμε τι είναι πιο σημαντικό. Να έχει υπερβολικό ειδικό βάρος η εκτελεστική εξουσία. Ήταν δύσκολο να προβούμε σε διορθώσεις. Γιατί? Αυτό το θέμα ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των κρατών, μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Αυτή η κατάσταση, αυτά τα παζάρια δείχνουν ότι η νομοθετική εξουσία πάντα είναι πιο αδύναμη ακόμη και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πριν από δύο μέρες, Πρόεδρε, είχαμε μία συνάντηση ε, με τον κύριο Λάντενμπουργκ για το θέμα της γειτονίας. Του κάναμε αυστηρές ερωτήσεις του είπαμε ότι οι παλιές διμερείς σχέσεις με τους γείτονες δεν έχουν αλλάξει και ότι δεν υπάρχουν νέες προτάσεις. Θα ήθελα να μας πείτε κύριε Αντιπρόεδρε, εσείς ως Τσεχική Προεδρία δίνετε μεγάλη σημασία στην γειτονία, στο θέμα της γειτονίας. Με ποια στοιχεία μπορείτε να προωθήσετε αυτή την πολιτική γειτονίας. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το θέμα της ενέργειας, το οποίο τέθηκε και από προλαλήσαντες. Πριν από δύο-τρεις μέρες, ασχοληθήκαμε με δύο εκθέσεις που προετοίμασαν οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, που είναι αρκετά αμφιλεγόμενες, που δείχνουν ότι υπάρχει μια μεγάλη πολεμική ανάμεσα στον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε, στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία, γιατί είναι πολύ δύσκολο να προγραμματίσουμε την ενεργειακή μας συνεργασία μακροπρόθεσμα και από την άλλη τι θα κάνουμε με όλους τους υπόλοιπους. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η προσέγγισή σας. Και το τελευταίο ερώτημα είναι το πρόβλημα της Τουρκίας. Γιατί το θέτω αυτό το ερώτημα. Για να επιλύσουμε τα προβλήματα της γειτονίας και να υπάρξει μια νέα όφηση σε αυτήν την πολιτική και για να προχωρήσουμε στον ενεργειακό τομέα, βλέπουμε μετά από αναλύσεις ότι η Τουρκία γίνεται ένα σημαντικός παράγοντας. Χωρίς ε, τη χώρα αυτή, χωρίς να υπάρξει μια σαφής δέσμευση από πλευράς ε, Τουρκίας, δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα ενεργειακά μας προβλήματα. Από την άλλη ξέρουμε ότι το μέλλον των αμοιβαίων σχέσεών μας είναι πολύ ζωφερό και σκοτεινό και ασαφές. Ποια είναι η προσέγγισή σας στο πρόβλημα αυτό με την Τουρκία. Uh, um, Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω ερωτήσεις που έθεσαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Αντιπρόεδρε, μια και μιλήσαμε για την επικύρωση της συνθήκης της, Λισαβόνας, ε, της Λισαβόνας στο Τσεχικό Κοινοβούλιο. Τα είχαμε συζητήσει τότε αυτά. Εσείς αναφέρατε δύο αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις. Θα μπορούσατε να εξηγήσετε λίγο καλύτερα ποια είναι αυτά τα δύο κείμενα στα οποία αναφερόσαστε. Ε, αναφερθήκατε και σε άλλες χώρες οι οποίες ε, ενίδησαν με τον ίδιο τρόπο. Ζητώ μια διευκρίνηση, δεν κατάλαβα περί την πρόκειται. Δεύτερον, δεν θέλω να επαναλάβω, αλλά να τονίσω τη σημασία κάποιων μεταβατικών λύσεων μια και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα βασίσουμε τις, ε, ευρωεκλογέ, τις ευρωεκλογές ή τις μελλοντικές μας δράσεις τους επόμενους μήνες μόνο στην Ίκαια, χωρίς να προετοιμαστούμε καθόλου για την ε, Λισαβόνα, η οποία είναι σε φάση επικύρωσης. Επομένως, χρειαζόμαστε μεταβατικές λύσεις. Θα πρέπει να προτείνουμε κάτι για τη σύνθεση του Κοινοβουλίου, αλλά χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας, δηλαδή της Προεδρίας. Επίσης, μιλήσατε για την επικοινωνία. Εμείς, από πλευράς Κοινοβουλίου, θέλουμε να υπάρχει συνεχής επικοινωνία και επικοινωνία με τους πολίτες. Αλλά να σε εμπιστήσω την προσοχή σε κάποια πράγματα που υπόθηκαν και χθες και σήμερα. Από τη μία θα πρέπει να μιλήσουμε στους πολίτες για την Ευρώπη. Γιατί κάποιοι από τους νόμους που έχουν προωθηθεί ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουν εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο, σε διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι, ευρωπαϊκά νομοθετήματα που δεν έχουν εφαρμοστεί. Για ποιο λόγο. Θα μπορούσε να το εξετάσει αυτό η Προεδρία και να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις. Πάντα για το θέμα της επικοινωνίας λέμε ότι θέλουμε οι πολίτες να εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά σε επίπεδο κρατών μελών η προπαγάνδα είναι πάντα εθνική, για τα εθνικά τεκτενόμενα. Αλλά δεν γίνεται κανένας λόγος για την ευρωπαϊκή διαδικασία, για τα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα. Αν δεν μπουν αυτά τα δύο θέματα, το εθνικό και το ευρωπαϊκό, στο ίδιο επίπεδο, το μήνυμά μας προς τους πολίτες ότι είναι πολύ όμορφο να ανήκει κανείς σε μια ευρωπαϊκή κοινότητα, αυτό το μήνυμα αποκλείεται να περάσει. Πάντα οι πολίτες θα είναι προσκολλημένοι στη δική τους εθνική κοινότητα και θα διαφορούν για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Πώς θα προσέλθουν λοιπόν μαζικά στις ευρωεκλογές αν δεν τους ενδιαφέρει η Ευρώπη. Τι θα μπορούσε να κάνει η Τσεχική Προεδρία πρακτικά για να ελκύσει τους πολίτες. Κύριε Βόντρα, κάποιες ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Παρακαλώ, μπορείτε να απαντήσετε. I like all the questions. <laughs> I hope you will like the answers. Μένα άρεσαν οι ερωτήσεις, λέει ο κύριος Βόντρα. Ελπίζω να σας αρέσουν και εσάς οι απαντήσεις μου. έχω ομαδοποιήσει τις ερωτήσεις. Θα απαντήσω σε κατηγορίες ερωτήσεων για να σας καλύψω όλους. Κύριε Πρόεδρε, εσείς ε, με ρωτήσατε τι είδους εγγύησεις μπορούμε να δώσουμε στην Ιρλανδία. Μας αναφέρατε κάποια άρθρα που διαβάσατε στο New Observer. Όλοι έχουμε διαβάσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Δεν έχει νόημα να τα ξαναπούμε αυτά. Η διατύπωση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι σαφής. Θα υπάρξει ένα follow-up για την εφαρμογή των συμπερασμάτων. Και βλέπω εγώ ότι η Προεδρία μας έχει να αντιμετωπίσει μία περίοδο που διαιρείται στα δύο. Τα θεσμικά θέματα θα εντατικοποιηθούν το δεύτερο διάστημα όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, τη δεύτερη περίοδο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν δεν θέλω να προδικάσω τις συζητήσεις που θα λάβουν χώρα τους επόμενους μήνες. Είμαστε μόλις στα μέσα Ιανουαρίου, είναι πολύ νωρίς. Πρέπει να τονίσουμε ότι η μορφή αυτών των ε, νομικών εγγυήσεων για την Ιρλανδία θα πρέπει να είναι αποδεκτή από όλα τα κράτη-μέλη. Αναφέρατε τον ε, πρόεδρο ε, της Τσεχικής Γερουσίας. Ήταν εδώ στις Βρυξέλλες να μιλήσει για το θέμα της διαφάνειας. Τον είδα πριν από δύο μέρες αλλά δεν είχα λάβει μέρος σε αυτή την ε, συνάντηση εγώ. Να σας αναφέρω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Οι απαραίτητες νομικές εγγύησεις θα δοθούν στα εξής τρία σημεία. Το πρώτο σημείο. Τίποτα στη συνθήκη της Λισαβόνας δεν θα αλλάξει ε, τίποτα για κανένα κράτος μέλος. Το τονίζω. Στο βαθμό που οι αρμοδιότητες, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την φορολογία. Ο Τσέχος γερουσιαστής απλώς α, ε, σας παρέπεμπε στα συμπεράσματα. Αυτό είναι τμήμα της πολιτικής συμφωνίας ε, που επετέφθη στις Βρυξέλλες το Δεκέμβριο με την παρουσία όλων των Ευρωπαίων ηγετών. Επίσης, μιλήσατε εν συντομία για τη Γάζα και τη Μέση Ανατολή. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει κάποια εργαλεία όντως για να αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα. Μας επιτρέπει να προβούμε σε μεγαλύτερο συντονισμό ε, μας δίνει λιγότερες ευκαιρίες να λέμε ο καθένας τα δικά του μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. για το φυσικό αέριο είχαμε κάποια περιθώρια ελιγμών. Εγώ αποφάσισα να πάω στο Κίεβο για να διαπραγματευτώ με τους Ουκρανούς και να τους πιέσω, ούτως ώστε να υπάρξει κάποια συμφωνία ε, για την ε, επιτήρηση του αγωγού φυσικού αερίου. Ο Ζαν Λιουκ Ντεάν έκανε κάποιες ερωτήσεις για το πώς θα επιλεγούν οι ευρωβουλευτές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα και περιμένουμε και τη δική σας συνεισφορά και την έκθεσή σας συγκεκριμένα. Φαντάζομαι θα την παρουσιάσετε αυτή την έκθεση τον Απρίλιο. Εδώ στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Θεωρώ ότι θα υπάρξει ευκαιρία να συναντηθούμε και να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Περιμένω να δω την έκθεσή σας. Το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο για κάποιες χώρες, το καταλαβαίνω αυτό. Και πιστεύω ότι τα μεταβατικά μέτρα σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η δήλωση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι σαφής για αυτό το θέμα. Υπάρχει μια πολιτική δέσμευση. Σε περίπτωση που τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, αυτή η δέσμευση θα πάρει και νομική μορφή. Αυτά τα μέτρα θα διαφοροποιήσουν τις διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα πρέπει να εφαρμοστεί και να υπάρξουν μάλλον ε, νομοθετήματα σε επίπεδο πρωτογενούς δικαίου. Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι όλα αυτά να εφαρμοστούν μέχρι το 2010. Έχουμε λοιπόν κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας. Επομένως, ε, δεν βρισκόμαστε κάπου στο κενό. Υπάρχει μια πολιτική δέσμευση από όλα τα κράτη-μέλη σε επίπεδο κρατών και κυβερνήσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολιτικό κενό και υπάρχει χρόνος να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Ε, τώρα, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον, την Πρόεδρο και το τι θα γίνει μετά τις εκλογές του Ιουνίου. Συμφωνήσαμε πάλι το Δεκέμβρη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε μια δήλωση που επισυνάπτεται στα συμπεράσματα πως για το ζήτημα του ορισμού του Πρόεδρου της ε, Κομισιόν θα ξεκινήσει αμέσως η ε, σχετική διαδικασία μετά τις ευρωεκλογέ. Νομίζω λοιπόν πως ο ρόλος μας είναι να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και να φτάσουμε σε μια πολιτική ε, συμφωνία. συγκεκριμένα για να οριστεί πρόεδρος ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο του Ιουνίου. Βεβαίως, σε κάθε φάση θα γίνουν σεβαστές οι διατάξεις της συνθήκης που θα ισχύει εκείνη τη στιγμή. Νομίζω είναι προφανές. Ο Ρίτσαρτ Κόρμπετ με ρώτησε ε, τι στοίχημα να παίξει. Ε, κοιτάξτε, πρέπει και εμένα να μου δώσετε γκανιώτα. Άμα είναι να σας δώσω συμβουλή για το στοίχημα. Πρέπει να το, το συμφωνήσουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει τώρα να σοβαρευτούμε. όπως σας είπα. Φαντάζομαι πως οι επιτροπές θα τελειώσουν το έργο τους ε, το Φεβρουάριο και μετά θα πάνε θα πάει το ζήτημα για ψηφοφορία στην Βουλή και μετά και στην ε, Γερουσία βεβαίως που απαιτείται πλουσία τριών πέμπτων το θέμα είναι στα χέρια των βουλευτών. Αλλά η κυβέρνηση εδώ έχει δεσμευτεί να προχωρήσει. Εγώ ψήφισα υπέρ. Είμαι και γερουσιαστής, γνωρίζω την ατμόσφαιρα στην γερουσία, ψηφίσω υπέρ και η ποιότητα της απόφασης είναι το σημαντικότερο. Είμαστε υπεύθυνη χώρα, αλλά πρέπει να γνωρίζετε πως είναι μια εσωτερική δημοκρατική διαδικασία οπότε οποιαδήποτε εξωτερική πίεση δεν νομίζω ότι βοηθάει. Αφήστε μας λοιπόν να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε μια δημοκρατική χώρα και υπεύθυνη χώρα. Νομίζω λοιπόν αυτοί οι δύο στόχοι, δηλαδή η δημοκρατία και η η υπευθυνότητα και τα, τα επίθετα αυτά, οι λέξεις αυτές αν θέλετε, είναι η απάντησή σας. και προς τον ε, Αντριάν Σεβερίν που ρώτησε τι εννοώ, ζήτησε διευκρινήσεις. κομμάτι της συνθήκης Λισαβόνας είναι αυτή η ρήτρα, η πασαρέλα, η λεγόμενη γέφυρα για την υιοθέτηση των ε, αλλαγών ε, στο σύστημα και κάποιες χώρες όταν ε, ψήφισαν τη συνθήκη της Λισαβόνας φρόντισαν να υπάρχει αυτή η λεγόμενη δημοκρατική εντολή, δηλαδή η κυβέρνηση να υποχρεούται να ζητήσει την συγκατάθεση του Κοινοβουλίου. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή και οι επιτροπές ε, εργάζονται σκληρά για να τα καταφέρουν έγκαιρα, οπότε δεν είναι νομίζω καμία δύσκολη υπόθεση, απλά θα τροποποιηθεί ο κανονισμός ε, του Κοινοβουλίου και των δύο σωμάτων. Λοιπόν, ο Άντριου Νταφ και ο Κάρλος Καρνέρο νομίζω ανέφεραν κάτι το οποίο δήλωσε ο Πρωθυπουργό ε, στο Κοινοβούλιο απαντώντας σε ερωτήσεις του ζητήθηκε μια διευκρίνηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ε, τύπου. Εν πάση περιπτώσει ήταν ένα τσεχικό αστείο η απάντησή του και δεν ξέρω αν μεταφράστηκε ή αν μεταφράζεται σωστά. Το αστείο Κοιτάξτε, υπάρχει κάποιο σκεπτικισμό από πλευρά Τσεχίας, αλλά αυτό δεν αφορά την ε, συνθήκη, αφορά την φύση της κοινωνίας. Έχοντας αντλήσει τα δάγματά μας από την ιστορία, να μελετήσετε την, την τσεχική ιστορία, πώς ξεκίνησε ετης πόλεμος με το τέλος της τσεχικής μεταρρύθμισης και με τη συμφωνία του μονάχου είναι λίγο διαφορετική η νοοτροπία και η ατμόσφαιρα με μια πρώην αυτοκρατορία όπως η Ισπανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο Έτσι διαμορφώνεται το κλίμα. Έτσι έχει το κλίμα. Ήταν ένα γνωστό τσεχικό αστείο που είναι... που λέει πώς πάμε φέτος, ε, χειρότερα από πέρσι και καλύτερα από του χρόνου. Είναι, εν πάση περιπτώσει, παροιμία στα τσέχικα. Είναι μια έκφραση. Αστείο ήταν λοιπόν και ο Πρωθυπουργός δήλωσε ξεκάθαρα πως ε, θα κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε και έχει ε, δεσμευτεί η κυβέρνηση να υποστηρίξει την συνθήκη και την επικύρωσή της. Και οπωσδήποτε δεν πρόκειται για τα θέμα της ποιότητας της ε, δημοκρατίας. Εάν δείτε τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία για την ε, μεταρρυθμιστική συνθήκη το 2007 έχουμε επενδύσει πάρα πολλά οι Τσέχοι διπλωμάτες μαζί με τους Ολλανδούς και κάποιους άλλους για να κάνουν την υπόθεση αυτή πιο διαφανή, να υπάρχει περισσότερος δημοκρατικός έλεγχος από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, δεν είναι θέμα λοιπόν δημοκρατίας. Είναι μάλλον θέμα επιρροής παρά δημοκρατίας. Αυτή είναι η εξήγηση. Αλλά νομίζω γνωρίζοντας την τσεχική νοοτροπία θα έλεγα πως πρέπει να παίξουμε έναν κάποιο ρόλο κατά διάρκεια της Προεδρίας μας και οπωσδήποτε τα δικά μας συμφέροντα είναι κοινά με τα δικά σας εδώ πέρα. Δηλαδή να διορθωθούν αυτά τα προβλήματα, να ενσωματωθεί και η Ιρλανδία, να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε όσο δυνατόν περισσότερους και να μην αποκλείσουμε κανέναν και είμαι πεπισμένος πως η Τσεχική Προεδρία μπορεί να παίξει εδώ ένα θετικό ρόλο σαν να βοηθήσει να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να φέρει ξανά και την Ιρλανδία εντός της συνθήκης γιατί πρέπει να είναι αποτέλεσμα έκφρασης της ελεύθερης ε, βούλησης και όχι να, να αναγκαστούν να παραδοθούν δηλαδή αφού τους στριμώξουμε. Ο Ενρίκε Μπαρόν Κρέσπο είπε κάτι για το εάν υπάρχει σχέση μεταξύ της ε, αντιπυραυλικής σπίδας και της ε, συνθήκης Λισαβόνας. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα αυτά. Ε, θα τα ψηφίσουμε εξχωριστά οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι πως ένα τμήμα του πολιτικού φάσματος, η κεντροαριστερά, έχει κάποιες αμφιβολίες για την ε, αντιπυραυλική ασπίδα και αναμένει τι θα πει η Αμερικανική κυβέρνηση ενώ στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος υπάρχουν κάποια ζητήματα για την ε, συνθήκη και υπάρχει βεβαίως και έτσι ατλαντισμός παραδοσιακός. Ποια είναι η λύση λοιπόν για εμάς ε, είναι μια ισορροπία. Χρειαζόμαστε και ευρωπαϊκές λύσεις και έναν ισχυρό υπερατλαντικό δεσμό σχέση. Δεν υπάρχει δηλαδή εδώ πέρα κάποια σύγκρουση ή κάποια αλυσίδα που συνδέει αυτά τα ζητήματα. Ε, the, the, the, the, elementary national consensus that και η, ε, η σχέση με την Ευρώπη και η σχέση με την Αμερική είναι πολύ σημαντική για μας. Τώρα από εκεί και πέρα ε, για την Τσεχική Προεδρία θα τα καταφέρουμε, ναι. Έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας σίγουρα η Προεδρία μας θα είναι διαφορετική από την προηγούμενη Προεδρία έχουμε διαφορετικές ικανότητες, διαφορετικές εμπειρίες θα είμαστε πιο μετριοπαθείς λέμε Ευρώπη χωρίς σύνορα αλλά αυτό δεν σημαίνει Ευρώπη χωρίς κανόνες και βεβαίως αυτό έτσι μια μετριοπαθή προεδρία μπορούμε να κάνουμε ούτως ή άλλως για να υπάρχει συνέχεια μεταξύ των προεδριών υπάρχει αυτό το πρόγραμμα των 18 μηνών και είμαστε σε επαφή και με τους Γάλλους φίλους και με τους Σουηδούς φίλους μπορείτε να δείτε και το κείμενο που περιγράφει αυτό το 18 μηνό πρόγραμμα και μπορείτε να δείτε ότι ακολουθούμε κάποια πολύ συγκεκριμένα ε, βήματα Τώρα για την μαζική προσέλευση των πολιτών στις εκλογές. Το είπαν κάμποση αυτό. Κοιτάξτε, για να είμαι τελείως ειλικρινής, από τις τελευταίες εκλογές τοπικές η πείρα μας ήταν ότι οι εκλογές αυτές είχαν μεγαλύτερες διαστάσεις τελικά δεν ήταν ούτε το, δεν ήταν τοπικές ακριβώς εκλογές, δημοτικές, περιφερειακές ήταν Ε, ε, για εθνικά ζητήματα έπαιξε ρόλο και η αντιπολίτευση βέβαια εκεί προωθών, προωθώντας μια κάποια νοοτροπία ε, τώρα μιλάμε για ευρωεκλογές υπάρχουν ευρωπαϊκά ζητήματα ε, ε πολύ ε, κάνουν δημοσκοπήσεις στο, στην κοινή γνώμη που λες εταιρείε που φτιάχνουν και μπύρες συγχλώρος και αφήσει αναφέρον ε, ερευνούν την κοινή γνώμη οπότε καταλαβαίνετε τι εννοώ και θα δούμε τι θα γίνει. of questions on a Τώρα ακούστηκαν και άλλα ε, θέματα ε, που κυρίως συζητούνται στην Επιτροπή Εξωτερικών Θεμάτων ε, ε, εταιρική σχέση με την Ανατολή βεβαίως τώρα η σχέση με τη Ρωσία το δεν ξέρω τι θα πρέπει να κάνουμε προηγούμενα που ε, προσπαθούσα να ανοίξω αυτό το μπουκάλι της Γκάσπρο τέλο πάντων και κόντεψε να εκραγεί ε, δεν πλήρωσα το το πλήρωσα το ότι δεν ήμουν αρκετά προσεκτικός Θα δούμε για τη Ρωσία τώρα για την Τουρκία ε, ίσως δεν είναι σκόπιμο να σας παρουσιάσω ούτε την προσωπική ούτε την εθνική μας άποψη. Να πω μοναχά ότι ένα θέμα είναι σημαντικό. Η, ενεργεια, η ασφάλεια εφοδιασμού ενέργειας είναι ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή και άρα η σχέση μας με την Τουρκία είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι ξεπέρασα το χρόνο μου, τον εξάντλησα. Ελπίζω να κάλυψα όλους. Σας ευχαριστώ. Yeah. Μάλιστα λέει ο πρόεδρος κύριε Αλεξάνδρ Φόντρα σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα παρεμπιπτόντως το νερό είναι από βελγική εταιρεία όχι ρώσικη εταιρεία Α, περιπτώσει νομίζω ότι ο διάλογος μαζί σας ήταν ε, ανοιχτός και ελεύθερος ε, μάθαμε κάποια πράγματα για την τσεχική προεδρία ε, πραγματικά θέλουμε να επιτύχει η προεδρία σας και η επιτροπή μας θα σας βοηθήσει ε, όσο μπορεί σας ευχαριστούμε που ήρθατε ελπίζουμε να σας ξαναδούμε ή να είστε σε στενή επαφή και με τους εισηγητές που ασχολούνται με θέματα σαν και αυτά που σας απασχολούν. Ευχαριστούμε πολύ. Στο επανειδήν.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 Συνεχίζουμε λοιπόν με τα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκεκριμένα το σημείο 9, προβλήματα και προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Η συγητής, ο κύριος Παναγιώτης Δημητρίου, Συνάδελφε Δημητρίου, σας ευχαριστούμε για την εργασία την οποία κάνετε. Υπάρχουν τέσσερις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και μετά θα ψηφι... και νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε τροπολογία 1 τώρα της κυρίας α όχι της κυρίας Σάτκοβα απεσύρθη τροπολογία 2 της κυρίας Σάτκοβα ποιος είναι υπέρ Δημήτριο. Dafür Εκθέση Δημητρίου υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Μποτόπουλος. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, Πάμε γρήγορα. Τροπολογία 5 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 Βοτόπουλος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τροπολογία 7 της κυρίας Τρακκόβα με μια προφορική τροπολογία είναι κανείς κατά τις προφορικές, Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και η τροπολογία 8 απεσύρθη και πάμε στην τελική ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ της έκθεσης Δημητρίου. Danke, wer ist Κατά. Αποχές. μια αποχή εγκρίνεται λοιπόν η έκθεση του κυρίου Δημητρίου. Συγχαρητήρια κύριε Δημητρίου. Σας ευχαριστούμε πολύ και παραμείνετε βεβαίω για να προχωρήσουμε και στις άλλες ψηφοφορίες. Σημείο 10. Ενεργός διάλογος με τους πολίτες σχετικά με την Ευρώπη. Η κυρία Κάουφμαν είναι η συγγήτρια. Ψηφοφορία. Τροπολογία 1 στράτκοβα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ ποιος είναι. Κατά. Uh, that was clear. Okay. Should be skeptical, like the Czech mentality. <laughs> Always be skeptical. So that is... Uh, λοιπόν, πρέπει να έχουμε και τις αμφιβολίες μας όπως και η τσεχική προεδρία. απορρίπτεται λοιπόν τροπολογία 2. Ευχαριστώ. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία υπέρ της έκθεσης Κάουφμαν, 3 Δεκαεφτά το σκορ εγκρίνεται η έκθεσή σας κυρία Κάουφμαν και σας ευχαριστούμε σημείο 11 της σημερινής σας διάδεξης ερμηνεία του άρθρου 149 του κανονισμού πρέπει να διευκρινίσουμε το πόσοι πρέπει να είναι, πόσοι βουλευτές πρέπει να είναι παρόντες για να μπορεί να ληφθεί απόφαση. Οι συντονιστές ε, το συζήτησαν το θέμα, απεδείχθη ότι δεν χρειάζεται έκθεση, απλώς μια επιστολή που πρέπει να σταλεί από τον πρόεδρο. Ε, έχετε την επιστολή, ποιος είναι υπέρ του κειμένου. Wer ist dagegen? Κατά. Αποχές. Δεκαέξι υπέρ ένας κατά μία αποχή. Το εκείνο που είναι το ενδιαφέρον είναι ότι υπήρξε μια αλλαγή το, σε σχέση με τον Ιούλιο έτσι ένα υπέρ έγινε κατά και ένα κατά είναι υπέρ τέλος πάντων Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη το 12 αναθεώρηση του κανονισμού σε σχέση με τη διαδικασία αναφορών Ζερά Ονέστα. Περνάμε στην Σοφορία, τροπολογία 22 Δημητρίου με μια προφορική τροπολογία του εισηγητή. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Ποιος είναι υπέρ λοιπόν. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στην τροπολογία 2 του εισηγητή ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 του εισηγητή με προφορική τροπολογία ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Ποιος... Κύριε Ονέστα. Cela concerne, vous savez, le... Ναι, Πρόεδρε, ε, εδώ μιλάμε για τον ελάχιστο αριθμό συναδέλφων στην Επιτροπή Αναφορών, ελάχιστο αριθμό που απαιτείται για να θεωρηθεί παραδεκτό ένα κείμενο. Ε, ένα τέταρτο της του συνολικού αριθμού της Επιτροπής. Αυτό είπαμε στην αρχή. Μετά άλλοι είπαν όχι, ένα τρίτο. Εγώ είμαι στη διάθεση της Επιτροπής, δεν έχω πρόβλημα και με ένα τρίτο και με ένα τέταρτο μπορώ να επιζήσω. Ε, αν νομίζετε ότι είναι βέβαια πολύ περίπλοκο ακολουθήστε τον κατάλογο ψηφοφορίας αλλά Ευχαριστώ χαιρετίζω τη φόρμουλα που βρήκε ο εισηγητής για να βγει από το αδιέξοδο. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν συνάδελφοι στη συζήτηση που είπαν ένα τέταρτο και τα λοιπά. Εμείς θέλουμε να επανέλθουμε στην άλλη ε, που είπαν ένα τρίτο εμείς θέλουμε να επανέλθουμε στην αρχική πρόταση του κυρίου Ονεστά στο ένα τέταρτο για να εδώ μιλάμε για τι, για το τι χρειάζεται για να μπει στην ημερήσια διάταξη αναφορά. Δεν μιλάμε για το περιεχόμενο είτε για συζήτηση του περιεχομένου. Για να μπει στην ημερήσια διάταξη μιλάμε και εγώ λέω ένα τέταρτο. Πρόεδρος, μα δεν νομίζω ότι υπάρχει ε, αντίρρηση σε αυτό. Ωραία λοιπόν, να προτείνουμε, να ψηφίσουμε λοιπόν το 4, την ανθρωπολογία ε, 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε οι άλλες καταπίπτουν. Για... Τώρα πάμε στο 27, ονεστά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 που είναι ταυτόσιμη με την 9 ή όχι. Αυτή δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. 11 11, τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ Α, απεσύρθη απεσύρθη πρόεδρε Antrag 20. 20 λοιπόν, τροπολογία 20 υπέρ. Υπέρ. Για την 20. Dagegen. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Και τελική ψηφοφορία τώρα για το σύνολο της έκθεσης Ονέστα υπέρ. Κατά Αποχές 20 υπέρ Μία ψήφος κατά Μία αποχή Συγχαρητήρια Θερμά κύριε Ονέστα ε, ε, Πάμε στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξη κατευθυντήριες γραμμές για μια πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της πρωτοβουλία πολιτών. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Κάουφμαν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πριν την ψηφοφορία να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους με τους οποίους τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες συνεργαστήκαμε επικοδομητικά, δηλαδή Λαμασούρ, Γκραμπόφσκα, Βιλουμπίτσκι, Φόγγεν, Χούμπερντάλ και να ευχαριστήσω και τον συναδελφό Κανέρο που συνέταξε τη γνωμοδότηση για την Επιτροπή Αναφορών. Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, είναι μια παράκληση προς την Γραμματεία να ρίξει μια ματιά ακόμα στην ε, διατύπωση. Στη μετάφραση νομίζω έγιναν κάποιες ανακρίβειες σε κάποιες γλώσσες. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Εκεί που λέγεται ε, εκεί που, που αναφέρω τη συνθήκη ε, βεβαίως έχω ξεκινήσει από τα γερμανικά. Στα αγγλικά όμως βλέπω πως ε, δεν πήραν το αγγλικό κείμενο της συνθήκης αλλά έγινε μετάφραση του δικό μου κειμένου. Π.χ. αυτό το οποίο λέγεται ε, απαιτεί από την Κομισιόν στα αγγλικά έγινε calls on ενώ είναι requests ε, στα αγγλικά το ζητά από την Κομισιόν. Το σε αυτό στην Κομισιόν. Οπότε θέλω να σας παρακαλώ εκεί όπου αναφέρεται η συνθήκη να κοιτάξετε το κείμενο της συνθήκης για να δείτε αν είναι σωστό σε όλες τις ε, γλώσσες. Ναι, σας ευχαριστώ. Εντάξει, είναι ένας μικρός μαραθώνιος, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ για την διαβούλευση που ήταν ευρύτατη, την είδα, ε, την έζησα. και πρόκειται βέβαια για μια πρόταση για να γίνει κάτι νόμος, οπότε έχει μεγάλη σημασία. Περνάμε στην ψηφοφορία συμβιβαστική τροπολογία 1 της εισηγήτριας που είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 της εισηγήτριας π 2 π P1 ήταν η πρώτη και τωρα π P2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά περνάμε στην τροπολογία DAF υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν είναι σίγουρη η γραμματεία, οπότε θα μετρήσουμε υπέρ της 36 του DAF. υπάρχει η πλειοψηφία για να λοιπόν. Τροπολογία 1 Τη ηγήτρια υπέρ. Κατά αποχέ. δεκτή. Τροπολογία 2 τη ηγήτρια υπέρ. Κατά αποχέ. δεκτή. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχέ. δεκτή. Τροπολογία 4 είναι συμβατή, οπότε περνάμε στην... Α, μπορεί άρα να ψηφιστεί. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές. Δεκτή. Τώρα περνάμε συμβαστική τροπολογία P3 υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές δεκτή. Τοπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τώρα περνάμε στην συμβιβαστική 1 της συγγήτριας υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συνεχίζουμε με την 11 Παπαστάμκου υπέρ κατά απορρίπτεται αποχές απορρίπτεται τροπολογία 12 υπέρ κατά πρέπει να ξαναμετρήσουμε ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 12 υπέρ αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ψηφίζουμε τώρα το αρχικό κείμενο του εκτιμώντας όμικρον υπέρ κατά απορρίπτεται. Τοπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε τώρα το αρχικό κείμενο Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεκτή. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 18 υπέρ Κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στην 19 με προφορική τροπολογία του κυρίου Δημητρίου. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά αποχές. Το ξανακάνουμε; Υπέρ της 20. 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ναι, παρακαλώ κυρία Κάφμαν. Δυστυχώς δεν με είδατε. Κατά την άποψή μου δεν έπρεπε να έχουμε ψηφίσει καν, γιατί είναι γλωσσικό το ζήτημα, αναφέρεται και στην ίδια την τροπολογία. Παρακαλώ να το ξαναδείτε. Και στην ε, άλλη, την 47 του κυρίου Δημητρίου, είναι επίσης γλωσσικό το ζήτημα που δεν αφορά τη γερμανική γλώσσα. Εκτός μικροφώνου ο πρόεδρος. Δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική P4 της εισηγήτριας ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές δεκτή.

Καταπίπτει. Όχι, δεν καταπίπτει γιατί δεν υιοθετήθηκε η 26. Οπότε πρέπει να ψηφίσουμε την 29. Η 29 υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται. Πολύ καλή αλλά απορρίπτεται. Συγγνώμη. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Α, να ελέγξουμε. Υπέρ λοιπόν. Αποχές. Ωραία. Ισοψηφία 9 με 9. Οπότε απορρίπτεται. Τριάντα ένα, λαμασού, ριπέρ. Μια στιγμούλα. Μου λένε τώρα πως ε, καλύπτεται αυτό στην συμβιβαστική 1. Όχι. Εντάξει, ψηφίζουμε την 31. Υπέρ της 31. κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην 34. Υπέρ. Κατά. υπέρ 9 κατά απορρίπτεται. Περνάμε Ναι, να το ξαναδούμε. Ποιος είναι υπέρ της 34 λάμα σου. εκεί. Κατά. Ο θαύματος τώρα είναι 11 με 9. Οπότε καμιά φορά αξίζει να, να ελέγξουμε. Ως εκθαύματος. Λοιπόν, συνεχίζουμε άρα με την 37. Καλύπτεται από τη συμβαστική 1. Because all but before. Yes, because we were already here. No. Yes. Okay. Äh, Kompromiss 1 hat äh, jetzt ab. Η συμβιβαστική 1 καλύπτει την 37 μέχρι τη 43 και περνάμε στις 44 Παπαστάμκου. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. αποχές δεκτή. 46. έξι ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 47 υπέρ. Γλωσσική. Είναι μόνο γλωσσική, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Ωραία. 48 υπέρ. κατά εποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή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 αποχές δεκτή 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εξήντα τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Εξήντα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ ναι. Κοιτάξτε, εφόσον η τροπολογία μου για διαγραφή όλου του παρατήματος έχει πάει σε πολλές τροπολογίες ζητώντας να διαγραφεί κομματάκι κομματάκι, εφόσον απορρίφθηκε η πρώτη, αποσύρω όλες τις υπόλοιπες, δηλαδή την 68, 71, 73, 75, 77 και 78 για να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Και το ίδιο νομίζω για τις 81, 82, 84, 86, 87 και την 93. Uh, <laughs> Αρκετές ε, τροπολογίες. Σας ευχαριστούμε που μας διευκολύνετε. Ναι, παρακαλώ. Κι εγώ σε αυτή την περίπτωση είμαι αναγκασμένος να διαγράψω, να αποσύρω δηλαδή την 69 και την 72. Αλλά την 74 θα ήθελα να την ψηφίσουμε και την 77 του κυρίου Κόρμπετ. Θα ήθελα να την ψηφίσουμε. 74 και 77 παραμένουν. 69 και 72 αποσύρονται. Επίσης παραμένει και 78. More. Άλλος κανείς. I accept Δέχομαι και άλλες προσφορές απόσυρσης advise me what was. We go now to 70 um, in favor. 70 υπέρ. Κατά. Εποχές. Κατά, άρα απορρίπτεται. Περνάμε στη... 74.

αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ογδόντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Wir sind dann schon 93 ήδη στην 93. Πάλι Κόρμπετ. Ποιο είναι υπέρ τη 93. Κατά. Αποχέ Απορρίφθηκε. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έχουν αποσυρθεί και αυτές οι τρεις Ρίτσαρντ. Οπότε ερχόμαστε στην συμβιβαστική 2 της ηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Οπότε περνάμε στην 103. 103. 103, 104, 105 έχουν αποσυρθεί. Ωραία. 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 107. Υπέρ κατά αποχές δεκτή 108 υπέρ κατά αποχές δεκτή 109 υπέρ κατά αποχές δεκτή για την γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών χρειαζόμαστε δύο ψηφοφορίες η πρόταση υπαριθμών 4, την οποία θα ψηφίσουμε τώρα και μετά το εκτιμώντας β. Πρώτα απ' όλα πρόταση 4, ποιος είναι υπέρ της Επιτροπής Αναφορών, κατά, αποχές απορρίπτεται, εκτιμώντας β, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία για την έκθεση Κάουφμαν υπέρ Ψηλά παρακαλώ τα χέρια. Αποχές. Οπότε η έκθεση εγκρίνεται με 15 έναντι 4. Συγχαρητήρια κυρία Κάφμαν για το έργο σας. Είχαμε μία και έχουμε μια σημαντική συζήτηση να κάνουμε με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους πολίτες. Και τώρα προχωρούμε στο σημείο 14 της ε, ημερήσιας διάταξης για τη δημόσια πρόσβαση στα, στα έγγραφα του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Η κυρία Γέτερμα εκεί είναι η συγγήτρια, τροπολογία 1 της συγγήτριας υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα για την τροπολογία 15 υπέρ. Τροπολογία 15 υπέρ.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 Dagegen. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τροπολογία 14 υπέρ. Dagegen. Κατά. Αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ποιος είναι υπέρ της έκθεσης στο σύνολό της. Κατά αποχές 20 ψήφοι υπέρ, μία κατά Πραγματικά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ευχαριστούμε για το έργο σας και φτάνουμε στα διάφορα στην ημερήσια διάταξη. Δεν έχω τίποτα εγώ στα διάφορα, οπότε σας δίνω... Α, Richard Corbett, σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης για τα πρακτικά, Πρόεδρε χτες είπατε ότι θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά εκτός αν γίνουν σχόλια μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Αν δεν κάνω λάθος υπήρξε κάποιο σχόλιο πρόεδρος. Όντως ο κύριος Ρίτσαρντ Κόρμπετ έχει πρόβλημα με τα πρακτικά της Επιτροπής Δευτέ της, ε, του Νοεμβρίου αμφισβητεί τη λίστα των παρισταμένων γιατί ο κύριος Μόουτ ήρθε, υπέγραψε αλλά δεν κάθισε στη θέση του, βγήκε κατευθείαν έξω από την αίθουσα. Αμφισβητεί λοιπόν του κατά πόσον ο κύριος Μόουτ συμμετέσχε στην συνεδρίαση. Νομίζω ότι ο κατάλογος παρουσιών θα πρέπει να αναφέρει ποιος έλαβε μέρος στην συνεδρίαση. Ε, έθεσα θέμα διαδικασίας. Το υπάρχει στα πρακτικά, αλλά η το διαδικαστικό αυτό ζήτημα έχει και μια συνέπεια να τροποποιηθεί η λίστα των παρισταμένων. Αυτή η συνέπεια δεν υλοποιήθηκε. Ο κύριος Μουτ. μια και εγώ είμαι ο λόγος αυτής της καταγγελίας που δημοσιεύτηκε στην Guardian την επόμενη μέρα δεν ξέρω μπορώ να φανταστώ πως θα ήθελα να πω στην Επιτροπή ότι ήμουν ασθενής εκείνη τη μέρα και δεν έλαβα μέρος σε τίποτα. Ζητώ συγγνώμη που σας ενοχλώ με προσωπικά μου ζητήματα. Ήρθα με κάθε καλή πρόθεση να συμμετάσχω στην Επιτροπή εκείνη τη μέρα αλλά αναγκάστηκα να φύγω και δεν μπόρεσα να ξανάρθω ζητώ συγγνώμη ε, με λυπούμε μάλλον που ο κύριος Κόρμπετ το θεωρεί αυτό απαράδεκτο αλλά νομίζω ότι δεν είμαι ο μόνος ούτε θα είμαι ο τελευταίος που του τυχαίνει κάτι τέτοιο έχει συμβεί και αλλού στο παρελθόν ευχαριστώ κολλήγη Κιόκοπ Uh, να διευκρινίσω κάτι. Είναι ένα σημαντικό θέμα, όχι μόνο για αυτή την Επιτροπή, αλλά για όλες τις Επιτροπές. Το θέμα της προσέλευσης ή όχι, ε, πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να συζητείτε ή όχι. Θα πρέπει να ζητήσουμε τεχνικές διευκρινήσεις, όχι μόνο από εσά πρόεδρε. Εσείς βεβαίως ελέγχετε τη δική σας συνεδρίαση, τη δική μας επιτροπή, αλλά το θέμα αυτό εκφεύγει από το πλαίσιο της Επιτροπής. Τι σημαίνει προσέλευση σε μια συνεδρίαση. Ε, τι σημαίνει μόνο ότι υπογράφω το Μητρό Παρισταμένων. Είναι κρίμα που τον κύριο Μόου τον έχουμε στυλιτεύσει. Μας εξήγησε την προσωπική του θέση, τα προσωπικά του προβλήματα, αλλά δεν είναι θέμα προσωπικό. Θα πρέπει να το διερευνήσουμε. Και εγώ θα ήθελα μια διευκρίνηση για το τι απαιτείται. Ε, αυτό αφορούσε ήδη από την αρχή της ε, συνεδρίασης. Ε, τι γίνεται αν συνεχίζεται η συνεδρίαση, κάποιος εμφανίστηκε για μία μικρή χρονική στιγμή και υπογράφει το μητρό παρισταμένο και φεύγει. Ε, μπορεί να έχει αποφασίσει ας πούμε ότι έχει κάτι πιο σημαντικό να κάνει. Ε, θεωρείται ότι έχει παραστεί στη συνεδρίαση, ότι έχει συμμετάσχει στη συνεδρίαση. θα ήθελα η γραμματεία να μας ενημερώσει και να συντονιστούμε λίγο και να το ψάξουμε το θέμα και με τις άλλες επιτροπές. Σωστό. Αυτό λέει ο πρόεδρος βέβαια εγώ δεν ήμουν παρών στη συνεδρίαση αυτή ήταν άλλος ο πρόεδρος αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει το θέμα και θα κάνω και μια συγκεκριμένη πρόταση ναι ε, ήθελα να τον δέσω εδώ στη συνεδρία του συνάδελφο Μότ αλλά δεν είχα σκηνή, δεν είχα σπάγκο λοιπόν κυρίες και κύριοι τώρα σοβαρά ε, εδώ τι προσπαθούμε να κάνουμε προσπαθούμε να ελέγξουμε οι μεν τους δε ε, στο, γίνεται μια προσπάθεια εδώ να πολιτικοποιηθούν κάποια πράγματα τα οποία ε, δεν θα έπρεπε να πολιτικοποιηθούν ξέρω κι εγώ από το παρελθόν ότι εξεμάνει εναντίον του συναδέλφου Μάρτιν ο οποίος ήταν ο μεγάλος ηθικολόγος ο οποίος όμως δεν ερχόταν ποτέ στις συνεδριάσεις και αλλά τελικά δεν έχει λόγο δεν νομίζω ότι έχουμε λόγο να αρχίσουμε τέτοιου είδους πολεμική εδώ, πολεμική ε, εδώ. Κοιτάξτε, σε τελευταία ανάλυση πότε είναι κανείς πράγματι παρόν και συμμετέχει στις συνεδρίες μετά από δύο λεπτά μετά την προσέλευσή του μετά από 30 λεπτά που βρίσκεται στη συνεδρίαση και δεν έχει λάβει μέρος γιατί μπορεί να πει κάποιος κοιμάται ή γιατί βαριέται ή γιατί δεν τον ενδιαφέρει δεν νομίζω ότι μπορούμε, μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση αυτά κάνω έκκληση λοιπόν να μην ε, ε, κάνουμε αυτού του είδους ε, έχουμε αυτού του είδους αντιπαραθέσεις εδώ στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ ο συνάδελφος Νταφ. Συμφωνώ. Και εγώ συχνά παραπονιέμαι για ανθρώπους που είναι στη συνεδρίαση ή δεν είναι στη συνεδρίαση. Ε, θα έλεγα να, να μην το συζητήσουμε περαιτέρω αυτό το θέμα. Ο κύριος Σονεστά. Δύο παρατηρήσεις. Το μητρό που υπάρχει στην αίθουσα είναι ένα μητρό για τους παρευρισκόμενους της Επιτροπής μας, αλλά και ε, στο Κοινοβούλιο. Γιατί για να πάρει κανείς το περδίεμ θα πρέπει να υπογράψει το μητρό, οπουδήποτε. Η υπογραφή σας εδώ δεν σημαίνει ότι είμαστε παρόντες μόνο στην Επιτροπή, αλλά δηλώνουμε ότι είμαστε παρόντες στο Κοινοβούλιο. Μπορούν οι συνάδελφοι να έρθουν λοιπόν να υπογράψουν και να φύγουν. Ε, δεν είναι υποχρεωμένοι να παραστούν στις ε, εργασίες της Επιτροπής, σημαίνει ότι είναι παρόντες στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το πρώτο. Στην τελευταία σύνοδο στο Στρασβούργο, ε, υπογράψαμε μία έκθεση με ένα ενδιαφέροντα τίτλο που λέει ότι τώρα και πριν από τις εκλογές θα καταστήσουμε δημόσιο το βαθμό προσέλευσης ε, στις Ολομέλειες και στις Επιτροπές. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό για τους συναδέλφους που θα είναι ξανά υποψήφοι. Εγώ δεν θα είμαι. Λοιπόν, προσοχή. Και ο Ρίτσαρτ τώρα που έθεσε το ζήτημα και μετά ο κ. Μαουτ δεν έγινε αυτό στην αρχή της ε, συνεδρίασης, κάπου στη μέση της συνεδρίασης έγινε. Ο εν λόγω βουλευτής μπήκε στην αίθουσα, υπέγραψε και αμέσως έφυγε. Πραγματικά είμαι στεναχωρημένος που, ακούμε, που ακούω ότι ήταν άρρωστος ο κύριος Μόουτ. Προφανώς του ήρθε απότομα. Τη στιγμή δηλαδή που υπέγραφε, του ήρθε ξαφνικά η αίσθηση αυτή, η ασθένεια αυτή. Ελπίζω να μην του ξανασυμβεί. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δεχόμαστε κατηγορίες στον τύπο α, για μέλη που έρχονται, υπογράφουν και δεν συμμετέχουν στις ε, διαδικασίες. Ε, είναι κρίμα κάτι τέτοιο. Ο κύριος Ονεστά είπε ότι αυτό το μητρό δείχνει ότι είμαστε παρόντες και στο Κοινοβούλιο. Δεν το αμφισβητώ προφανώς ήταν στο Κοινοβούλιο, ε, ταξίδεψε, υπέγραψε για να δηλώσει ότι είναι παρόν στο Κοινοβούλιο. Το Μητρό ισχύει και γι' αυτό. Αλλά για τα πρακτικά της δικής μας συνεδρίασης δεν θα πρέπει να θεωρείται ο κύριος Μόουτ παρόν. Γιατί δεν συμμετείχε στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να τον θεωρούμε λοιπόν παρόντα. Και μια και τέθηκε ως διαδικαστικό τη στιγμή της συνεδρίασης, καταγράφτηκε στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης και επομένως είναι παράδοξο που το Μητρό των Παρευρισκομένων στο τέλος συνεδρίασης αναφέρει ακόμα αυτό το όνομα, παρότι τέθηκε θέμα. Και είπαμε ότι δεν παρίσταται ο κύριος Μόουτ. Κύριος Μόουτ. Τι να σας πω, τα έχω χάσει σχεδόν. Το γεγονός και μόνο ότι κάθομαι εδώ και ακούω ότι έφτασα αργά ε, και πρέπει να εξηγήσω ότι το αεροπλάνο μου έφτασε αργά ή ότι δεν αισθάνθηκα καλά και ήρθα για να υπογράψω. Ήρθα γιατί προφανώς ήθελα να συμμετάσχω στις εργασίες επιτροπής, αλλά δεν μπόρεσα, όπως αποδείχτηκε. Σε ό,τι αφορά τη λέξη συμμετοχή, πολλές φορές κάποιοι βουλευτές, ίσως όχι ο κ. Κόρμπετ, ε, παρίσταντο, αλλά δεν συμμετείχαν κατά ανάγκη στις ε, συζητήσεις. Χτες ε, είχαμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Ο κ. Άλιστερ ήρθε, υπέγραψε, έκανε μια σύντομη δήλωση και μετά πήγε στην Επιτροπή Ελίας. Γιατί τον ενδιέφερε ένα συγκεκριμένο θέμα ε, και χρειάστηκε να μιλήσει κιόλα για αυτό το θέμα. Τον επέκριναν γιατί δεν ε, παρέμεινε για να ακούσει τα σοφά λόγια του κυρίου Κόρμπετ. Φαντάζομαι θα διαβάσω τα τεκτενόμενα αυτού του τμήματος της συνεδρίασης ε, στην αυριανή Guardian, στο Diary. Εγώ, όπως σας εξήγησα, ήθελα να συμμετάσχω σε αυτή τη συνεδρίαση, αλλά δεν μπόρεσα τελικά. Ωραία, λέει ο πρόεδρος. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμη η συζήτηση. Ο ο κύριος να ζητεί το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο γιατί νομίζω ότι τα πρακτικά έτσι όπως φτιάχτηκαν είναι σωστά. διο επιβεβαιώνει όχι μόνο όχι τη συμμετοχή ε, του Ευρωβουλευτή αλλά την παρουσία το το γεγονός ότι μπήκε σε ένα κατάλογο παρισταμένων. Αυτό επιβεβαιώνουν τα πρακτικά πρόεδρος, είδατε οι νομικοί, είδατε πάντα βρίσκουν μια ερμηνεία χρήσιμη και καλή. Λοιπόν μετά από αυτά που είπε ο κύριος Σονεστά και ο κύριος Λένε δεν τροποποιούμε τα πρακτικά και δεν πρόκειται να αρχίσουμε ε, πολεμική εδώ για το πότε συμμετέχει κανείς και πότε όχι. Πέρα στις συνεδρίες μπορείτε να φύγετε όλοι τώρα.